Λοιπόν, συνάδελφοι, όσοι θέλετε να αποχωρήσετε παρακαλώ ταχαίως και ησύχως. Περνάμε τώρα στην ε, εξήγηση των ε, ψήφων. Έχω διαφόρους εγγεγραμμένους στον κατάλογο. Charles Γκόρεντς, πρώτος.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 Αυτή η μέθοδος ε, θα πρέπει να αφορά όλα τα κοινοτικά όργανα και όλα τα κράτη-μέλη ε, στα πλαίσια της διαδικασίας λήψης αποφάσεως και αυτό από το αρχικό στάδιο. Ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε την ε, χρηματοοικονομική κρίση το 2008 από την ομάδα των τεσσάρων κυρίως ήταν αντίθετη με αυτήν την μέθοδο που ανέφερε και χθε το απόγευμα ο κύριος Μπαρόζο. Το 2008 επιματέω Α, περιμέναμε να επαναφέρει στην τάξη τα πράγματα ο κύριος Μπαρόζο η Ευρωπαϊκή Ένωση η Γαλλία το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία η Ιταλία, τα μέλη του Σωμάτας των Τεσσάρων δεν είναι α, μόνα τους υπάρχουν όλα τα υπόλοιπα κρατημένη τα οποία δεν συμμετέσχαν στην σημαντική αυτή φάση της διαδικασίας λήψης αποφάσεων το 2008. Οπότε με τα λόγια σας, ε, Πρόεδρε Μπαρόζο, δεν τιμάτε την διαδικασία που εσείς ο ίδιος πρεσβεύετε. Γι' αυτό δεν μπορώ να υποστηρίξω την ε, εκλογή σας. Ζητώ συγγνώμη κύριε Πρόεδρε, αλλά είναι πολύ, δύσκολο να μιλήσει κανείς ε, με όλο αυτό εδώ το θόρυβο. Ευχαριστώ. Επαναλαμβάνω, όσοι θέλετε να αποχωρήσετε παρακαλώ αποχωρήσατε ταχαίως και ησύχως. Ο κύριος Ριβαλίνη παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε μετά την ε, παρέμφασή μου θα πω και δύο λόγια στα ναπολετάνικα. Όχι για φολοκλωρικούς λόγους, αλλά για να προσελκύσω την προσοχή των ε, μέσων ενημέρωσης. Πρόεδρε Μπαρόζο, σας υπερψήφισα και ελπίζω να είστε πρόεδρος όλης της Ευρώπης, ακόμα και της Νότιας Ιταλίας, που είναι η πόρτα εισόδου στην Ευρώπη. Στο σταυροδρόμι μεταξύ των Υπήρων και με μια κουλτούρα φιλοξενίας εξαιρετικά σημαντικό για όλη τη γυραιά Ευρώπη, την γυραιά Ήπειρο. Και τώρα που αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, η Ευρώπη θα πρέπει να παρέμβει υποστηρίζοντας τον νότο της Ιταλίας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 Ξέρω ότι είσαστε νέος κύριε, αλλά για την επόμενη φορά ένα λεπτό παρακαλώ. Επεξηγήσεις ψήφου ένα λεπτό. Ο επόμενος ομιλητής είναι ο κύριος Ντάνιελ Χάνεν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ίσως ο χρόνος μας συνήθισε στις ιεροτελεστίες τις οποίες μόλις βιώσαμε, αλλά ε, είναι είναι, ε, ε, βλέπετε όμως πόσο σημαντικό είναι να υπάρχει εις ε, τα χέρια μίας μη άμεσα εκλεγμένης ε, ε η εκλογή του Προέδρου. Ε, λοιπόν, δεν έχω προσωπικά προβλήματα με τον Χωσέ Μανουέλ Μπαρόζο. Ε, εφόσον αυτόν θέλει το κοινοβούλιο ας είναι αυτός και όχι κάποιος άλλος από ότι ε, ένας Άγγλος ε, πολιτικός τον οποίο δεν συμπαθώ καθόλου αλλά το σύστημα αυτό δίδει στα, σε νομοθέτες τους οποίους δεν εκλέγουμε άμεθα τη δυνατότητα να νομοθετούν. Ευχαριστώ κύριος Καμάλ. Αντίθετα με τον συνάδελφο που μίλησε προηγουμένω, θα πω ότι και εγώ επιφυλάξει είχα για τον κύριο Μπαρό για να ξαναεκλεχθεί πρόεδρο Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ε, είναι δεσμευμένο ε, για την περαιτέρω ολοκλήρωση παρά τη βούληση των λαών τη Ευρώπη. Ε, στην συνεδρίαση των Ευρωπαίων Συντηρητικών μα μας είπε ότι είναι υπέρ τη εφιού νομοθεσία. Μα τι σημαίνει αυτό. Οι πολίτε θεωρούν ότι ε, η έλλειψη νομοθεσία δεν συνιστά εν πάση περιπτώσει ευφυή νομοθεσία και αν είναι υπέρ αυτού πρέπει να μεριμνήσει ώστε σε κάθε οδηγία να κάνει ε, μια ικανή αξιολόγηση αντικτύπου Ευρωπαϊκή Επιτροπή του χρόνου έχουμε παραδείγματο χάρη θα έχουμε την οδηγία για τα εναλλακτικά επενδυτικά ταμεία. Δεν έχει κάνει μελέτη οικονομικού αντικτύπου η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λέει δεν γίνεται. Μα υπό αυτές τις συνθήκες πώς θα είναι η φιέστερη νομοθεσία που ψηφίζουμε. Ας το ξανασκεφτεί ο κύριος Μπάρος. Ευχαριστώ. Thank you. Now I have Mr. Ευχαριστούμε. Ο κύριος Άντριου Μπρον για ένα λεπτό. To oppose the joint uh, motion for resolution on forest fires αντιτάχθηκαν στο κοινό ψήφισμα για τις δασικές ε, πυρκαγιές παρόλο που συμφωνώ οι ευρωπαϊκές χώρες εθελοντικά να συνεργάζονται για να καταπολεμούν τις ε, πυρκαγιές και τις συνέπειες αυτών. Αλλά αντιτίθεμαι με οποιαδήποτε δημιουργία ε, οργάνων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο που θα ασκούν πίεση στις εθνικές κυβερνήσεις για θέματα που δεν είναι αρμοδιότητά τους. Εφιστώ την προσοχή στα τμήματα 03, 07 και 08 του κοινοψηφίσματος. Οι διατάξεις αυτές ε, ανθρωπιστική απόκριση στην, ε, στις ε, καταστάσεις που δημιουργηθήκαν και είναι ένα βήμα για τη δημιουργία του Europe Aid όπως λέει η έκθεση Μπάνι. Ευχαριστώ. And finally, Mr. Και τέλος ο κύριος Κλέης. Eh, Ευχαριστώ πρόεδρε. Απόσχα κατά την ε, ψηφοφορία για το ψήφισμα διότι ταλανίζομαι από αμφιβολίες και ανησυχίες. Είναι πολύ καλές οι προθέσεις του ψηφίσματος ενδυνάμωση της ε, πολιτικής προστασίας, ανταλλαγής εμπειρογνωμόνων, μεθόδων εργασίας, ε, είδαμε δασικές πυρκαγιές ε, το περασμένο καλοκαίρι που έλαβαν τέτοιες διαστάσεις ε, που καθιστούν την συνεργασία απόλυτα απαραίτητη. Αλλά αυτή η συνεργασία ήδη λαμβάνει η χώρα μεταξύ των κρατών μελών. Και δεν λέω ότι δεν μπορεί να εμβαθυνθεί, να εμβαθυνθεί αλλά δεν έχει καμία χρησιμότητα, καμία προστιθέμενη αξία η δημιουργία ενός ιδιαίτερου σώματος. Μία γραφειοκρατική δομή θα δημιουργήσουμε ε, που θα δημιουργήσει προσκόμματα στη συνεργασία που ήδη έχουν τα κράτη-μέλη. Άλλος της επιθυμεί να λάβει το λόγο για να επεξηγήσει την ψήφο του ή την ψήφο της. Όχι. Διακόπτουμε καλή όρεξη. Θα τα ξαναπούμε στις 3.